Now, is it fixed? Is it okay? Yes. Now it's okay. Thank you. Thank you. Now apparently it's working. So let's let's make it smooth. I was saying, we have. Έλεγα λέει ο πρόεδρος ότι έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ συγχρόνως με την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ που είστε παρόντες, που θυσιάσατε την Ολομέλεια και σε εργαστούμε γρήγορα. Έχουμε ψηφοφορίες και γι' αυτό παρακαλώ να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες έτοιμες γιατί θα ψηφίσουμε. Έχουμε δύο ψηφοφορίες. Δεύτερη ψηφοφορία. Υπάρχει σύμφωνα με το άρθρο 214 μία απόφαση των συντονιστών, τις οποίες έχουν αμφισβητήσει Πράγμα που σημαίνει συγκεκριμένη περίπτωση ότι Ζητείτε από την ECR να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση, μία οργανώσης που ενεργούν στην ε, Καταλωνία τίθεται σε αμφισβήτηση. Οι συντονιστέ έχουν διαφορετική άποψη. Θα την ψηφίσουμε για να δούμε αν ναι ή όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο δεύτερο, η δεύτερη ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα, θα ψηφίσουμε για το κύριο θέμα μα, που είναι η ψηφοφορία για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Χθε είδαμε του υποψηφίου. Έχουμε τρεις ε, υποψηφίους, καλύπτονται ε, γλώσσες πάρα πολλές εκτός ε, από, τα εστονικά, τα κροατικά και τα δανέζικα τα έχουμε παθητικά. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού θα πρέπει για τον ε, Ευρωπαίο Επόπτη να υπάρχει κοινή συμφωνία, όχι συνένεση, κοινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εάν όχι, θα ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Έχουμε ήδη δει μια τέτοιου είδου κατάσταση, αλλά πρώτα απ' όλα να δούμε αν υπάρχει κοινή συμφωνία για του υποψηφίου για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν και ονομαστική ψηφοφορία και ηλεκτρονική. Έχετε τα τρία κουμπάκια, το ναι, το όχι και τις εποχές. Το κουμπάκι στα αριστερά θα είναι για να ψηφίσετε τον κύριο Έρνετ Ζάμπο. Το μεσαίο κουμπάκι τον κύριο Βόισικ Βιβορόφσκι. Και το δεξί κουμπάκι για τον Γιάν Πάντοβα. Το καταλάβατε? Αριστερά Σάμπο, στη μέση Βιβορόφσκι. Πάντοβα στα δεξιά να είστε βέβαιοι ότι θα ψηφίσετε το σωστό κουμπάκι σύμφωνα με αυτό που επιθυμείτε. Σε περίπτωση που έχουμε δύο επικρατέστερους με πάρα πολύ ε, μικρή διαφορά, θα ξαναψηφίσουμε μεταξύ των υποψηφίων αυτών για να δούμε ποιον προτιμούμε. Και αυτά τα αποτελέσματα θα δοθούν στην διάσκεψη των Προέδρων και αν ενδεχομένω θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία. Διαφορετικά, η πλειοψηφία των ε, εκφραζόμενων ψήφων θα είναι αυτή που θα αποτελέσει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Goal. Ψηφίσατε όλοι. Υπάρχει ένας παραπάνω συνάδελφος στο ΕΛΚ. Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα έχουμε τον ακριβή ρυθμό. Λίγη η ψηφοφορία. How did it go? It's, I understand it's three to the right. Λοιπόν, 3 Σάμπο, 25 Πάντοβα, 36 Βιμπορόσκι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Εδώ έχουμε την επιστολή για την ε, συνδιάσκεψη των Προέδρων και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να αναφέρουμε δηλαδή το αποτέλεσμα της ψηφοφορία αυτής για να έχουμε κοινή συμφωνία με το Συμβούλιο. Τώρα για την ψηφοφορία κατόπιν ετήματος ECR. Διαδικαστικό είναι αυτό που θέλετε. Δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας, απλά το διαβάσατε. Δεν το είδαμε. γιατί δεν το είδαμε σε κάποια οθόνη. Ναι, ήταν σαφές το αποτέλεσμα της ψηφοφορία, ε, ψηφοφορίας, λέει ο Πρόεδρος. Το πρώτο ήταν ο κύριος Ζιβορόσκι, δύο Πάντοβα και το τρία ήταν ε, ο κύριος Ζάμπο. Και εκεί τελειώνει η υπόθεση. Έχουμε κι εμείς ένα διαδικαστικό για το επόμενο θέμα. Ποιος το υποβάλλει το διαδικαστικό αυτό θέμα. Εσείς, κυρία Ρίβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλαμε να καταγγείλουμε ότι το Vox τορπιλίζει την κανονική, την ομαλή διαδικασία της Επιτροπής και τη δουλειά των συντονιστών. Ε, ζητώ να υπάρχει σεβασμός στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι συντονιστές και, και οι θεσμικοί φορείς. Στην Καταλωνία δεν υπάρχει καμία ε, ε, τρομοκρατική οπλισμένη ομάδα που να ονομάζεται CDR, CDR. Υπάρχει ένας φορέας που έχει υποστηριχθεί από τη Διεθνή Αμνηστία και άλλους διεθνείς φορείς. Μιλούμε για διαδηλώσεις και διακοπές της κυκλοφορίας ε, των οδικών αξώνων, αλλά όχι η τρομοκρατική δραστηριότητα. Μιλούμε για τους γείτονέ μας, μιλούμε για κανονικούς ανθρώπους που διαδηλώνουν. Ε, κυρία Ρίβα, με όλο το σεβασμό, όταν ζητάτε επιδιαδικαστικού, ε, πρέπει να αναφέρεστε σε άρθρο του κανονισμού που να άπτεται διαδικασίας, όχι για να κάνετε δήλωση πολιτική επί της ουσία. este voto decir sí, nuestro punto de vista. No, no, sí, sí, ha, ha disfrutado de un minuto para exponer su punto de vista, pero solo sugiero que cuando se levante la mano, I'm, I'm only suggesting that when it comes to a point of order, when it comes to a point of order, you actually make a point of order, which is called... Τώρα ξαναακούμε τον Πρόεδρο που μιλάει για το διαδικαστικό. Πρέπει, για το διαδικαστικό μιλούμε επί της διαδικασίας, όχι επί της ουσίας δεν ζητούμε το λόγο επί διαδικαστικού για να κάνουμε πολιτική δήλωση, λέω. Συμφωνείτε. Κύριε Θαρθαλέχο, ε, επί διαδικαστικού, εκτός μικροφώνου ο ομιλητής. Αλλά, λέει ο ομιλητής, συνεχίζει, να μην μετατρέψουμε το θέμα σε συζήτηση επί της ουσίας. Υπάρχει έρευνα όμως επί από τις αρμόδιες αρχές στην Ισπανία, ήθελα πλέον να πω. Εκτός μικροφώνου. Vote. Let's vote. Because we I mean, we a clear cut. Ας ψηφίσουμε γιατί εδώ έχουμε σαφή ψηφοφορία. Σύσταση των συντονιστών να απορρίψουμε την πρόταση του ECR. Το ECR δικαιούται να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία. Δικαιούται. Και θα ψηφίσουμε. Επομένως, όσοι από εσάς υποστηρίζουν την πρόταση των συντονιστών να μην συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στη διάταξη, να ψηφίσουν συν. Αυτοί που διαφωνούν με την σύσταση των συντονιστών και συμφωνούν με το ECR να ψηφίσουν πλην. Έχουμε δύο δυνατότητες εδώ πέρα της αποχής. Συν και πλην. Εντάξει. Κυρία Κανκό, ε, επιδιαδικαστικού Ερώτηση, Πρόεδρε. Σε αυτό το πράγμα πώς θα ψηφίσω συν και πλήν, ε, Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Το συν είναι το αριστερό κουμπάκι και το πλήν ε, είναι το δεξί κουμπάκι. Αλλά όχι το μεσαίο, το μεσαίο είναι η αποχή. Συν στα αριστερά, πλην στα δεξιά. Αποχή στο μέσον. Ωραία. Τώρα λοιπόν ψηφίζομαι. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρασε. Ενεκρίθη η σύσταση των συντονιστών και τέλος για το θέμα αυτό. Και τέλος γενικά, αλλά να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 2 Δεκεμβρίου. Από τις 3 το απόγευμα. Την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας μέρα.